Ερχόμαστε τώρα στη διάταξη των εργασιών. Σύμφωνα με το άρθρο 137 ε, ενέκρινε η διάσκεψη των Προέδρων στις 18 του μηνός στην οριστική τελική ε, ημερήσια διάταξη, το σχέδιο μάλλον, ε, και δεν υπάρχει καμία διαφωνία, οπότε και αποφασίζεται έτσι η διάταξη των εργασιών, όπως ορίστηκε στο τελικό σχέδιο ημερήσιας διάταξης. Πριν